226 παράγραφο 4 ε, θα θεωρηθούν οι ερμηνείες αυτές ως εγκριθήσεις. Και τώρα προχωρούμε στην τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Ε, Για τη σημερινή ημέρα δεν έχω προτάσεις τροποποίησης ε, με βάση το άρθρο 194 και με βάση την, το, το κείμενο της τελικής ημερήσιας διάταξης. Ούτε για αύριο έχω προτάσεις αλλαγής. Για το είναι Τετάρτη ε, υπάρχει πρόταση σε σχέση με την αλλαγή της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις ε, με το Νοοθετικό Συμβούλιο το Παλαιστινιακό να αναφερθεί ε, το να αναβληθεί η συνάντηση αυτή για να ε, γίνουν οι απαραίτητε διαβουλεύσει. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα, θα ήθελα να κάνουμε μια παρατήρηση. Ε, αν ψηφίσουμε για την πρόταση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί αναπομπή του θέματος στη διάσκεψη των Προέδρων με την παράκληση το θέμα αυτό να τύχει διαβούλευση με την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Για την πρόταση ζητεί το λόγο ο κύριος Πρέντα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μόλις ε, αναφέρατε και εσείς και εμείς θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση είναι άκρο σημαντική. Πριν από την Ολομέλεια θα πρέπει να γίνει ε, μία ανταλλαγή απόψεων στην ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, γιατί η ΑΦΕΤ δεν έχει επί του παρόντος ασχοληθεί με αυτό το θέμα και θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέντα. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο υπέρ της πρότασης, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Α, όχι, κανείς. Ο κύριος εγώ κύριε Πρόεδρε θα μιλήσω εναντίον κύριε Πρόεδρε όπως αναφερθήκετε με βάση τον κανονισμό ε, είναι η Ολομέλεια που αποφασίζει για την αλλαγή του ονόματος στις αντιπροσωπείες μετά από εισήγηση της διάσκεψης των Προέδρων και εδώ έχουμε εισήγηση από τη διάσκεψη των Προέδρων άρα θεωρώ ότι με βάση τον κανονισμό πρέπει να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ε, ε, δεν θα ήθελα να μπω επί της ουσίας αλλά είναι γνωστό ότι από το 2013 σε όλο το εύρος των σχέσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τον όρο Παλαιστίνη και όχι η Παλαιστινιακή Αρχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Είναι σαφές το αίτημα, μιλάμε για την αναπομπή στην διάσκεψη των Προέδρων του θέματος για να διαβουλευτεί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων το θέμα. Όποιος είναι υπέρ της πρότασης της κυρίου Πρέντα, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Υπέρ της πρότασης του κυρίου Πρέντα. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το αίτημα. Νομίζω ότι ήταν σαφής η πλειοψηφία. Εντάξει. Αν θέλετε, ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Haben alle Abgeordneten. Ψήφισαν όλοι οι βουλευτές. Να περιμένω, να περιμένω λίγο, ακόμα μην ανησυχείτε καθόλου. Ερωτώ ξανά. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Μάλιστα. Πέρασε τη ψηφοφορία λοιπόν. 152 υπέρ, 180 κατά, απορρίπτεται το αίτημα, 42 αποχές. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν θα παραμείνει όσο είχε προτεθεί. Το ΕΛΚ ζητά μετά τη δήλωση της ΥΠΑ της για την κατάσταση στη Λευκορωσία να καταρτιστεί ψήφισμα και να ολοκληρωθούν διαβουλεύσεις για το ψήφισμα. Ο κύριος Πρέντα θα πάρει το λόγο για να αιτιολογήσει το αίτημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να έχω μεγαλύτερη επιτυχία με τη Λευκορωσία. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μία χρονική στιγμή όπου θα πρέπει να έχουμε συνενετική θέση σε επίπεδο κοινοβουλίου, όχι μόνο για την ανταλλαγή απόψεων. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε τη θέση μας επί ενός ε, κειμένου το οποίο υποστηρίζουν οι πολιτικές μας ομάδες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Θα ήθελε κανείς να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο του κυρίου Πρέντα. Όχι. Θέλει να πάρει κανείς το λόγο κατά του αιτήματο. Όχι. Α. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ο κύριος Μαρνίκενς. Πρόεδρε. Δεν ε, πιστεύω ότι πρέπει να βιαστούμε. Είναι πραγματικά πρόωρο να περάσει ένα τέτοιο ψήφισμα, γιατί τώρα βρισκόμαστε σε μια τεράστια κρίση προσφύγων. Μπορούμε να συζητήσουμε το ψήφισμα αυτό μια διαφορετική χρονική στιγμή, σε μια διαφορετική ολομέλεια. Good. Der Antrag von Herrn Preda ε, Μάλιστα. Λευκορωσία με ψήφισμα. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματος του κυρίου Πρέντα. Ποιος είναι κατά της πρότασης του κυρίου Πρέντα. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Χρειάζεται τώρα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρας. Ψήφισαν 204 υπέρ, 169 κατά, 7 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η πρόταση. So, jetzt müssen Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν ε, θα πρέπει να πάρετε τα μολύβια στο χέρι γιατί θα πρέπει να σας πω τι προκύπτει με τροποποιημένη ε, ημερήσια διάταξη. Ψήφισμα. Αύριο είναι η προθεσμία, 8 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα το πρωί. Λίγη η προθεσμία για το ψήφισμα. Για τροπολογίες και ε, κοινά ψηφίσματα την ε, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10 για τροπολογίες στα κοινά ψηφίσματα την ε, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 11 η ώρα. Η προθεσμία. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις προβλεπόμενες ώρες ψηφοφορίας. Για την Τετάρτη η ομάδα των Πρασίνων ζητάει δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΕΠΑΤΗ εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία για την κατάσταση στην Τουρκία και ζητούν να συνοδευτεί από ψήφισμα την Τετάρτη το απόγευμα όλα αυτά. Η ψηφοφορία για το ψήφισμα θέλουν να λάβει χώρα στην επόμενη, στη δεύτερη του Σεπτεμβρίου. Η κυρία Χάρμς έχει το λόγο για να τη λογίσει την πρόταση αυτή. Πρόεδρε, αξιότιμη συναδελφή, από τότε που συζητήσαμε την έκθεση προόδου για την Τουρκία και την ψηφίσαμε και από τις εκλογές στην Τουρκία έχουν συμβεί πάρα πολλά στη χώρα αυτή. Πολλοί έχουν καλωσορίσει την εκλογή της ε, κυβέρνηση Ερντογάν και την καταπολέμηση του ίσης. Αλλά παράλληλα υπήρχαν και πολύ αρνητικέ εξελίξεις στην Τουρκία. Η ειρηνευτική διαδικασία με τους ε, Κούρδους ε, τερματίστηκε. Η δίωξη δημοσιογράφων και άλλων προσώπων που είναι αντίθετα προς το καθεστώ συνεχίζεται με εντυπωσιακό ρυθμό και Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι μάλιστα, εξωτερικοί ανταποκριτές ε, διώκονται ως τρομοκράτες. Σήμερα το πρωί έγινε δίωξη στην Χουριέτ, τη μεγάλη όμιλο στην Τουρκία που αντίκειται στο καθεστώς. Και νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να απαιτήσουμε την κυρία Μογερίνη να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Γιατί αφενός θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στην Τουρκία η κυβέρνηση Ερντογάν για λόγους και σκοπιμότητες εξουσίας ρίχνει την χώρα στο παρελθόν και εκ παραλλήλου ανησυχούμε για την κατάσταση με τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα πρέπει να ανησυχούμε και να φροντίσουμε και για το ενιαίο μέτωπο κατά του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν που μας οθούν να ζητήσουμε από την κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ, διακόπτη ο Πρόεδρος. Ο Ποιος θέλει να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο της κυρίας Χάρμας, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα έχει να προσθέσει κανείς τα όσα έχει πει η συνάδελφος, γιατί πράγματι η Τουρκία βρίσκεται σε μια έκρηθμη κατάσταση έχουμε μια εξέλιξη συγκρούσεων και πολέμων σχεδόν σε όλα τα μέτωπα που έχουν να κάνουν με τα σύνορα της Τουρκίας και πολύ περισσότερο μια σύγκρουση με τους Κούρδους, επαναφορά της αιματηρής υπόθεσης προηγούμενων ετών ε, με πολύ μεγάλους κινδύνους για όλους τους πολίτες της Τουρκίας αλλά δυστυχώς και για όλους τους λαούς της περιφέρειας. Υπογραμμίζω και εγώ ότι δυστυχώς όλη αυτή η υπόθεση εξελίσσεται γιατί ο κύριος Ερτογάν θέλει μέσα από την ανασφάλεια που δημιουργείται στους Τούρκους πολίτες σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση να στραφούν ξανά υπέρ του κόμματος του. Και είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό πρώτα απ' όλα να μην το βλέπει κανείς και δεύτερο το Κοινοβούλιο να μην έρθει σε μια συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα, να καταθέσει την άποψή του και να σπρώξει τον κύριο Ερτογάν προς τη σωστή κατεύθυνση, αν αυτό είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο κατά της πρότασης αυτής. Ο κύριος Φερχόφστατ ζήτησε διαδικαστικό. Για άλλο ζήτημα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Πρέντα, λοιπόν, να πάρει το λόγο κατά της πρότασης. Απλώς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι είμαστε κατά αυτής της ιδέας ε, για μια συζήτηση για την Τουρκία αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή πρόκειται για μια συγκεκριμένη πολιτική θέση ε, αυτής, αυτού του κόμματος και το θέμα της μετανάστευσης και των τρομοκρατών θα συζητηθεί σε άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δεν θα ήταν σκόπιμο να μπούμε σε μια ε, πολιτολογία ε, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την άκρα αριστερά και την Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να ψηφίσουμε σχετικά με την πρόταση αυτή, την πρόταση της κυρίας Χάρμς για μία δήλωση της Αντιπροέδρου με ψήφισμα. Ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διατάξη για ποιος είναι υπέρ της πρότασης αυτής παρακαλώ. Υπέρ της πρότασης της κυρίας Χάρμς. Κατά. Αποχές. Ναι, αλλά μου δεν σηκώνετε τα χέρια σας, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς να ξέρω τι ψηφίζετε. Σας παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Να ελέγξουμε τότε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, παρακαλώ. Πέρας ψηφορίας, παρακαλώ. 153 οι ψήφοι υπέρ, 180 οι ψήφοι κατά, 36 αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Φερχόφστατ τώρα ζήτησε το λόγο για την Τετάρτη. Πρόεδρε, όπως ξέρετε, είχα ζητήσει την παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη συζήτησή μας ε, την Τετάρτη για την ε, μετανάστευση, όχι για την κατάσταση της Ένωσης για την μετανάστευση, γιατί πιστεύω ότι είναι ουσιώδες και απαραίτητο σε μια τέτοια κρίση που διανύουμε να είναι εδώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου για να συζητήσει την κρίση αυτή. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέα πρόταση. Το πρόβλημα όμω δεν είναι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ενιαίο μέτωπο που ψήφισε το ψήφισμα τον Απρίλιο. Το πρόβλημα είναι το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη που δεν επιδεικνύουν ενιαίο μέτωπο και αλληλεγγύη στο θέμα αυτό και για το λόγο λοιπόν ζητώ εκ νέου ο Στάσκ, Τάσκ μετά από προσωπικό σας αίτημα να παραστεί την Τετάρτη το πρωί στη συζήτηση για τη μετανάστευση. Κύριε Φερχόφστατ, μετά τη διάσκεψη των Προέδρων, το θέμα το έδωσα και στο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χωρίς όμως να έχω λάβει μέχρι τώρα θετική απάντηση. Μετά τη σημερινή συνεδρίαση θα τηλεφωνήσω στον πρόεδρο άλλη μια φορά. Ε, ναι, τουλάχιστον από μ, ορισμένους από την Ολομέλεια. Όχι ομόφωνα. Ε, δείξτε μου εμπιστοσύνη ε, ότι θα, μπορέ, θα το πω στον πρόεδρο ότι θεωρώ ότι θα είναι το καλό να παρευρίσκεται. Λοιπόν, δεν ζητεί κανεί το λόγο για την Τετάρτη, για την Πέμπτη δεν έχω ε, αιτήματα για τροποποιήσεις. Με την εξαίρεση της παρατήρησης για την ημερήσια διάταξη του συναδέλφου